Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. La séance est reprise. Κυρίσω την επανέναρξη των εργασιών της Επιτροπής μας. Επιβεβαιώνω ότι η κυρία Γεωργίεβα θα έλθει στην Επιτροπή μας αύριο το πρωί. 11 συγκεκριμένα το πρωί για να μας παρουσιάσει τη δεσμή μέτρων που αποφάσισε η Επιτροπή με θέμα την πολιτική και τις απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις σε σχέση με το μεταναστευτικό. Σε ό,τι αφορά τη μέση διάταξη, τώρα θέλω να σας ενημερώσω ότι μετά την εξέταση και την ψήφιση της έκθεσης 8 θα εξετάσουμε την έκθεση 8α της κυρίας ε, Γκάρτσια Θάμπαλ για τον ε, διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 6 του 2015. Συνεχίζουμε την εξέταση των τροπολογιών. Από εκεί που αφήσαμε το θέμα την προηγούμενη ε, βραδιά, δηλαδή κατηγορία 4. Δύο μπλοκ από συμβιβασμούς έχουμε καταρχάς δύο δέσμες. Πρώτη υποδέσμη, πρώτο sub-block για την αποκατάσταση. Ποιοι είστε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω κάποιον να απέχει. Εγκρίνεται αυτή η συμβαστική πρόταση. Δεύτερο υπό μπλοκ. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και η αυτή υποδέσμη. Και περνάμε στις χωριστές ψηφοφορίες. Έχουμε μια σειρά τροπολογιών το 010302, η τροπολογία ΑΓΚΟ 7257, μπάτς 4392, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται, μάλλον απορρίπτονται οι δύο τροπολογίες, η FTD 7983 ψηφίζουμε, ψήφι ΠΕΡ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 0103-06 γραμμή, η FTT 7984, τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα. 4415 ψήφι υπέρ. Κατά. Όχι, ε, κατά, ναι. Αποχές. Απορρίπτεται. 05-05-04-02, μπατ 44-14. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στο ίδιο κονδύλιο EFDD 79-78 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται, 1903-01-01, μπάτζ 44-71, υπέρ, κατά, αποχές, 19, 1903 1903-01-02, γραμμή. Δύο τροπολογίες, μπάτζ 44-72, μπάτζ 44-73, ψήφι κατά αποχές απορρίπτονται 19.03.01.03 δύο τροπολές badge 44.74 badge 44.75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 19.03.01.05 γραμμή badge 44.78 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε, 19.03.01.06 badge 44.79 ψήφι κατά αποχές απορρίψετε. 19.03.01.07 και S10 4.000 η τροπολογία badge 43.08 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19.03.01.07 Τροπολογία EFTD 79.80 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 19.06.01 μπάτ 44.84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19.06.01 Badge 43.29 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 21.02.04 γκουε 73.24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21.02.05 ENF 81.26 ψήφι Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 21.06.02 ENF 81.28 ψήφι Κατά αποχές απορρίπτεται. 22.02.03.01 γραμμή. EFTD 79-76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22-02-03-02. Η τροπολογία EFDD 79-77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 04 04 Μπάτζ 45-84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19.02.01 η τροπολογία 74, ε, συγγνώμη, 44.69 μπάτζ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στην ίδια γραμμή μπάτζ 40.56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19.02.02 Badge 4481 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19.03.01.06 Άλντε 80.64 Badge 42.24 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ Έχετε βάλει τις κάρτες στο μηχάνημα. Άρχεται ψηφοφορία. 16 υπέρ 14 κατά δύο εποχές εγκρίνεται, εγκρίνονται. 19.03.07 Μπάτζ 40.52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η διαγραμμή Μπάτζ 40.72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19.03.02 Μπάτζ 40.55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στη 19.04.01 μπάτζ 44.84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στη 19.05.01 μπάτζ 40.47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην 20.02.01 Badge 4065 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21.02.01 Τροπολογίες. 3 στον αριθμό. ΦΑΜ 6022. Γκου 7323. Badge 4486. Ψήφι υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται την τροπολογία. 16 ψήφοι κατά και 14 υπέρ. Και είχαμε και δύο αποχές. Πηγαίνουμε στις παρατηρήσεις. 21.02.02 μπάζ 40.45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21.02.03 η badge 40.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην 21.02.04 ΔΕΒΕ 57.05 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπάτζε 4230 του κ. Ρούμπιχ. Είναι ταυτός καλύπτεται. Η Μπάτζ 4046 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην 21.02.05 ΔΕΒΕ 57.06 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η μπάτζ 46-37 ταυτόσιμη καλύπτεται άρα μπάτζ 40-43 ψήφι πέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην 21-02-07-03 καταρχάς η ντεβε 57-10 ψήφι πέρ κατά αποχές εγκρίνεται η μπάτζ 42-31 καλύπτεται και πηγαίνουμε στην αλλη 80 80-84 και στην μπάτζ 40-36 ταυτόσιμες α καλύπτονται μπάτζ 41-13 ψηφίζουμε ψήφι πέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Όχι. 21.02.07.05 ΔΕΒΕ 57.12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21.02.51.04 η μπάτζ 41.45 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται στην 210401 η badge 4048 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται στην 210501 υπέρ λέει ο πρόεδρος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η τροπολογία. 22.02.03.01 Badge 4058 υπέρ κατά αποχές δεν σηκώνετε τα χέρια γι' αυτό θα ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται τροπολογία, αλλά παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. 25.04.01.01 μπατ 40.54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22.04.01.03 Μπατζ 42.61 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22.04.02. Άλντε 80.82. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρα το ίδιο και η badge 4297. Πάμε στην badge 4264. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 22-04-02-03, η τροπολογία ALDE 80-73, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Η μπάτζη 42-98 καλύπτεται. Στη γραμμή 23-01-06-01, μπάτζ 41-44, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές Απορρίπτεται. Στην 23.02.01 η ΔΕΒ 57.19 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. S&D 7140 είναι ταυτόσημη, εγκρίνεται, καλύπτεται τέλος πάντων. Η ΑΦΕΤ 5121 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με την κατηγορία 4. Alors, les députés sont Bien. Un changement technique. Τεχνική φύσεω αλλαγή έγινε όσον αφορά τον κατάλογο που έχετε στη διάθεσή σα. Ο νέο κατάλογο διανέμεται τώρα. Ο κ. Γενικό Εισηγητή μα επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τεχνική αλλαγή και όχι κάτι ουσιαστικό. Αφορά τι πληρωμέ. κατάλογο των πιλωτικών προγραμμάτων, προπαρασκευαστικών δράσεων. Έχετε όλοι το έγγραφο. Θα μπορέσω λοιπόν να το ψηφίσουμε, να το θέσω σε ψηφοφορία. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν υπάρχουν. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ο κατάλογος εγκρίνεται. Πάμε στα άλλα, σας κατηγορίες, στα άλλα τμήματα, δίνω το λόγο, στον συγκεκριτή, τον Ζεράχ Ντεπρέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, δεν φανταζόμουν ότι θα είχα ευθύνη των άλλων τμήματων, ότι θα ήταν τόσο μεγάλη περιπέτεια όπως αυτή που έζησα. Να ευχαριστήσω τις άλλες πολιτικές ομάδες όσον αφορά τη συνεργασία τους για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι πριν το καλοκαίρι είχαμε συμφωνήσει κάτι που εγκρίθηκε και από την Ολομέλεια, να προτείνουμε ένα προπολογισμό αυξημένο του Κοινοβουλίου κατά 1,6% όσον αφορά τις τρέχους δαπάνες, συν 15 εκατομμύρια έκτακτες δαπάνες, κυρίως τα τμήματα ασφαλείας των κτηρίων και ασφαλεία στον κυβερνοχώρο. Τα νέα γεγονότα συνέβησαν μετά τη δημιουργία μιας πολιτικής ομάδας, οπότε επιληφθήκαμε τριών τροπολογιών. Ε, δύο δεν είχαν σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά τον προπολογισμό, πάνω από τη εκατομμύρια δημιουργία νέων θέσεων προς όφελο. Ε, της νέας ομάδας και 3,5 εκατομμύρια για διάφορες συμβάσεις ε, για τις πολιτικές ομάδες. Αυξήθηκαν οι πιστώσεις κατά 6 εκατομμύρια 702.000 ε, με τη συνεργασία των άλλων πολιτικών ομάδων και υπό την πίεση μίας από αυτές τις πολιτικές ομάδες αποφασίστηκε και καταφέραμε να αντισταθμίσουμε πλήρως την αύξηση των πιστώσεων. Ο προπολογισμό του Κοινοβουλίου, ο οποίος έχει υποβληθεί τώρα, ε, υπόψη αυτές τις αντισταθμίσεις ε, και είναι αυτά που είχαμε πριν το πριν το καλοκαίρι 1,6% αύξηση κανονικέ κανονικές δαπάνε δαπάνες του Κοινοβουλίου και 15 εκατομμύρια για τις έκτακτες δαπάνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες συνεργασία τους ακόμα και αν ο συμβιβασμό δεν δεν αντικατοπίζει πλήρω τι απόψει μου και αυτό που θα ήθελα. Όσον αφορά τα άλλα τμήματα και κατηγορίε, τα σε αυτά σε άλλη ευκαιρία. Εν γέννη, κάνω δύο εξαιρέσει. Εν γέννη, προτείνω να αποκατασταθούν οι πιστώσει που είχαν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δύο εξαιρέσει. Η πρώτη είναι το ε, δικαστήριο, διότι θα πρέπει να έχει περισσότερα μέσα το δικαστήριο, διότι αυξήθηκε ο αριθμό των δικαστών και αυτή η αύξηση του αριθμού των δικαστών συνεπάγεται και αύξηση των διοικητικών δυνατοτήτων, άρα να αποκατασταθεί προτείνω ο προπολογισμό επιστώσει που είχαν ζητηθεί από το δικαστήριο, διότι θεωρώ ότι οι δαπάνε αυτέ είναι απόλυτα δικαιολογημένε που ετούνται. Υπάρχει δεύτερη αλλαγή που προτείνω. Ε, γνωρίζω ότι η πόρα που έχει από την επιτύχει η και αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Επαναλαμβάνω η επιλογή που έκανα και που θα επέμενα σε αυτή ακόμα και αν παραμείνω μόνος μου είναι να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράση. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επίτροπης πρότεινε αύξηση των πιστώσεων 5,1% αύξηση. Το Συμβούλιο από την πλευρά του έδινε μια αύξηση 3,79%. Ε, έκανα τις δέωσες αναλύσεις δεν θα αναφέρω τι αναλύσει. Ανέλησα όλε τι αιτήσει και πιστώσει και κατέξω συμπέρασμα, ο, και αυτό είναι ο συμβιβασμό που σα προτείνεται, να κάνουμε το εξή. Πρώτον, να επιβεβαιώσουμε όσον αφορά την ασφάλεια διαβίβαση πληροφοριών και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την κρυπτογράφηση στοιχείων, να επιβεβαιώσουμε τι πιστώσει που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τι εγκρίνουμε για άλλες ε, κατηγορίες και ένα παράδειγμα θα δώσω όσον αφορά κάποιες άλλα, άλλα κονδύλια Υπάρχει μεγάλη απόκληση εκτίμηση μεταξύ του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποφάσισα να βγάλω το μέσο όρο μεταξύ των δύο. Εν γέννη να προτείνω μια αύξηση 4,6% εκεί που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά 5,1% και το Συμβούλιο έδινε 3,79%. Διευκρινίζω λοιπόν ότι αν ήταν να ακολουθήσουμε την πρόταση που ε, υποβάλλω, οι πιστώσει που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα αυξηθούν κατά 4,6%. Γιατί έκανα συμβιβασμό σε κάποια δεδομένη στιγμή, κυρίω όσον αφορά τα κτίρια κλπ. Διότι διαπίστωσα, παραδείγματο χάρη, ότι όσον αφορά τη θέση για τα κτίρια και σχετικέ δαπάνε, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών υπήρξε μια αύξηση ουσιαστικά κατά 70 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε οι πιστώσει σχετικέ με τα κτίρια αυξήθηκαν, διπλασιάστηκαν πρακτικά κατά τη διάρκεια τη τελευταία τριετία. Δεν είμαι πεπισμένο λοιπόν ότι στι παρούσε περιστάσει η πολιτική των επενδύσεων στον αφορά τα κτίρια αποτελεί μια προτεραιότητα απόλυτη τη Ένωση. Επιβεβαιώνω και γι' αυτό επιβεβαιώνω ότι εγώ στηρίζω τη συμβαστική πρόταση που σας έχω υποβάλει. Επαναλαμβάνω, δεν τιμωρώ κανένα, προτείνω μια αύξηση 4,1% και σε κάποιες περιπτώσεις δεν εστερίζω το τύπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι θεωρώ κυρίως στον τομέα αυτών οι αυξήσει των πιστώσεων είναι αδικαιολόγητε ε, και άσκοπε σε αυτή τη φάση. Έχω δεύτερη τροπολογία που αποτέλεσε αντικείμενο μια ε, επίμαχη συζητήσεω να βάλουμε στο αποθεματικό κάποιες πιστώσεις, αλλά αυτά δεν τα βάλα στο συμβιβασμό, προτείνω αυτά να ψηφιστούν ξεχωριστά. Πρώτη, να βάλω στο αποθεματικό τι πιστώσει που ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και κάτι που στήριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το άνοιγμα μέσα στην προσωπή στο Ιράν. Να βάλουμε στο αποθεματικό δεν σημαίνει ότι οι πιστώσει δεν είναι διαθέσιμε. Είναι στο κονδύλι, είναι στη γραμμή. Δεν αρνούμε το να μια αντιπροσωπεία στο Ιράν. Πιστεύω δύο πράγματα όμω. Το πρώτο είναι ότι όταν έχουμε να κάνουμε μια δικτατορία κατά τη γνώση μου, δεν είναι μεγάλη δημοκρατία το Ιράν, δεν είναι δημοκρατία, έχουμε κάθε λόγο ε, να είμαστε πιο διστακτικοί, πιο συνετοί από ότι όταν έχουμε σε, έχουμε σε επαφή με μια δημοκρατία διαπιστωμένη. Και δεύτερον, οι όροι που θέτω για να έρθει ε, να ελευθερωθεί το απόθεμα είναι κάτι δικαιολογημένο. Ε, το Ιράν να σεβαστεί τι δεσμεύσει τι οποίε ανέλαβε στη συμφωνία που συνήθι τον Ιούλιο και που κυρώθηκε από όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ότι η Διεθνή Υπηρεσία Ατομική Ενεργεία θα έχει διαπιστώσει και θα έχει εξακριβώσει ότι το Ιράν έχει σταματήσει κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση ε, χρήσεω πυρηνική ενέργεια σε στρατιωτικού σκοπού και αυτό θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με του όρου συμφωνία κατά τη διάρκεια του 2016. Εγώ δεν είμαι αντίθετο στο να ανοίξει με αντιπροσωπεία στο Ιράν. Λέω απλώ ότι ζητώ να υπάρξει μια απόδειξη ότι κινούνται καλή την πίστη οι Ιρανικέ αρχέ στον τομέα. Και δεν θα ήθελα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση κατά την οποία σε κάποια στιγμή θα έχουμε ανοίξει μια αντιπροσωπεία ενώ η Διεθνή Υπηρεσία Ατομική Ενεργεία θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το Ιράν δεν έχει σεβαστεί τι δεσμεύσει και να λάβει. Αυτό που προτείνω λοιπόν εδώ είναι ένας τρόπος να ασκήσουμε πιέσεις στις Ιρανικές αρχές, ούτως ώστε να σεβαστούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και αυτές που προβλέπονται από την συνηθίσια συμφωνία. Ειδού κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω, αυτά ήθελα να τονίσω. Ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία τους που με στήριξαν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερος ε, το Γενικό Εισηγητή για τα άλλα τμήματα. Εκεί η συνεργασία υπήρξε σχεδόν τέλεια και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, συνεργάτες, κυρίως τη γραμματεία της Επιτροπής Προπολογισμών για την εξαιρετική δουλειά που έκανε, καθώς και τους συνεργάτες της ομάδας και τους προσωπικούς μου συνεργάτες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και με τα χαράς ε, θα περιμένω να με κρίνετε. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ όλους εκείνους και εκείνες που σας συνόδευσαν στο όλο εγχείρημα. Χαιρετίζω λοιπόν τις προσπάθειες που, την αυταπάρνησή σας και τις προσπάθειες που καταβάλατε. Εκφράζω τη χαρά μου ότι χάρη, διότι χάρη σε εσάς ε, έχουμε αντισταθμίσει τις ε, έκτακτες δαπάνες που αφορούσαν τη δημιουργία μιας ε, καινούργιας ομάδας και αυξημένες δαπάνες επίσης που αφορούσαν τις αμοιβέ των συμβασιούχων που εργάζονται για την ομάδα θα ήθελα να πω τώρα εντελώ προσωπικά ότι οι αρχέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι αρμόδιε για τα δημοσιονομικά, εξαρτώνται κατά πολύ από την υποδειγματική εργασία και την αυστηρότητα που δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Προπολογισμών πάνω σε αυτό έχει κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει. Ε, θα επανέλθω σίγουρα επ' αυτής της κατευθύνσεως, επ' αυτού του στοιχείου κάνατε το εφικτόν επιδιώκοντας συμβιβασμό και έχω κάθε επίγνωση ότι ε, έπρεπε να δείξετε μια αυταπάρνηση ώστε να καταλήξετε σε αυτά τα συμπεράσματα. Τούτο λεχθέντος λοιπόν θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Ρούμπιχ επιθυμεί να πει κάτι. Μάλιστα, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία. Νομίζω καταλήξαμε σε έναν θετικό συμβιβασμό στον προϋπολογισμό. Μένουμε κάτω από το 20% της κατηγορίας 5. Πολύ ξεκάθαρο αυτό, ενώ την προηγούμενη φορά δεν ήταν τόσο εύκολο να κάνουμε αυτό το βήμα πρόοδου. Έχουμε λοιπόν καταθέσει έναν λιτό προϋπολογισμό. Είναι σημαντικό αυτό. Ενισχύουμε ταυτόχρονα τη δημοκρατία στο ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας νέους, προσφέροντας νέες θέσεις στη νέα πολιτική ομάδα, προσφέρουμε τα μέσα που χρειάζονται για την εργασία τους στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό αυτό το αίτημα για μας. Και ο διευθυντής στη νέα πολιτική ομάδα μπαίνει σε κατηγορία βιστολογική Α14. Βλέπω ότι, θεωρώ δηλαδή ότι πρόκειται για ένα βήμα μπροστά και ενίσχυση των πολιτικών ομάδων στην ε, δημοκρατία, στην ευρωπαϊκή δημοκρατία. Τώρα, δεύτερο, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εδώ έχουμε το πρόβλημα, η αναβάθμιση των δικαστών στον κατά επιδίω δηλαδή, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα γι' αυτό νομική βάση. Περιμέναμε πρώτα οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές να δημιουργήσουν την απαραίτητη νομική βάση και γι' αυτό θα χρειαστεί να διαμορφωθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Για να μην προκαταλάβουμε το έργο των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, το ίδιο λέγω για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Εκεί η Επιτροπή Εξωτερικών τοποθετήθηκε ξεκάθαρα για την αντιπροσωπεία στο Ιράν, χωρίς μάλιστα να προβλέψει αποθεματικό. Και με την κατάσταση κρίσεως στην Ιεμένη, αλλά και για τη συνεργασία με την ε, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Παρακολούθηση των Πυρηνικών Όπλων πρέπει να μπορούμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Εκεί δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε με τον ε, εισηγητή ούτε και η πολιτική ομάδα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση επί τόπου να μπορεί να συμμετέχει και στις προσπάθειες που γίνονται. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προσφέρει υποστήριξη στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να διαμορφωθεί και να ε, τοποθετηθεί αμέσως η αντιπροσωπή αυτή. Σημαντικό μέρος των συγκρούσεων που βλέπουμε στην περιοχή αυτού του κόσμου προέρχεται από εκείνη την περιοχή. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η θέση μας και θα τοποθετηθούμε κατά της θέσεως του εισηγητή. Εν τέλει θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε θαυμάσια μαζί μας. Και ευχαριστώ όλες και όλους που συνεργάστηκαν μαζί μας, μας ενημέρωσαν ορθά και είμαι εν τέλει πεπισμένος ότι η ψηφοφορία θα αποδώσει καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Μήπως υπάρχει κάποιος συνάδελφος το λόγο, δεν βλέπω να υπάρχει. Οπότε περνάμε στην ψηφοφορία. Καταρχάς τη γενική στρατηγική του εισηγητή, δηλαδή να αποκατασταθεί το σχέδιο προπολογισμού, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Ψηφίστηκε αυτό. Τμήμα 2, κατηγορία 2. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο. Ομαδική ψηφοφορία, όλο το μπλοκ. Όσον αφορά τις τροπολογίες 79, 58, 79, 57, 79, 59 60, 61, 62, 63, 64, 65. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι τροπολογίες αυτές απορρίπτονται. Για τα αποθεματικό για τη γραμμή 2000, τροπολογία των πρασίνων 7709 και προπολογισμο 4512 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτονται. Κατηγορία 4 του δικαστήριου. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες 2200, 2202, 2203, 2205 υπέρ. Κατά. Άποχες. Και αυτή η ομάδα των τροπολογιών εγκρίνεται για το αποθεματικό στη γραμμή 1000 Μπότ 4311 της κυρίας Γκρέσλε υπέρ. Η κυρία Γκράσλιν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπότζ 12, υπέρ. Κατά. Θα διεξαχθεί έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος που ξεκινάει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 17 ψήφοι υπέρ, 15 ψήφοι κατά. Μποτ 43-15 υπέρ κατά άποχες απορρίπτονται. πρόταση εισηγητού όσον αφορά την κατηγορία 6, τμήμα 6, η ESC, e, γραμμές S6, S1, BODS 2401 και στη γραμμή 1220 BODS 2402 μαζί τα ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται ξεχωριστές τα ψηφορίες. Γραμμή 1400 EFTD 7987 ξεχωριστές ψηφορίες. Λοιπόν, μετά 79, 88, 79, 89, 90, 79, 91, 92, όλες μαζί, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Στις άλλες παρατηρήσεις, στη γραμμή 1004, Bodge 4605 per κατά, αποχές, απορρίπτεται. η προτάσεις του για την κατηγορία 7, το τμήμα 7, Ψηφίζουμε μαζί τις τροπολογίες 2500, 508, 2501, 2502, 2503, 2505, 2506, 2507, 2509, 2510, 2500 υπέρ. Κατά. Άποχες. Αυτές οι τροπολογίες εγκρίνονται. Έχουμε τώρα άλλες ομαδικές Τροπολογίες EFTD 7996, 7995, 7997, 7998, 7999. ...251, 252, 253, 254 και 255 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτονται αυτές οι τροπολογίες. Για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις μάλλον, στη γραμμή 1000 Bots 4490 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται αυτή η τροπολογία. Προτάσεις του εισηγητού για το τμήμα 10, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Έχουμε σειρά τροπολογιών. Μπότζ 2803, 2800, 2801, 2803. 2803 προφορική τροπολογία του συγητή σειρά τροπολογιών προφορικών 2803 ψηφίζουμε όλες μαζί αυτές τις τροπολογίες ποιος είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτονται αυτές οι τροπολογίες. Τροπολογίες που θα ψηφιστούν μαζί σε μπλοκ, σε ομάδα, μπορούν να ψηφιστούν. Διότι δεν υιοθετήθηκαν τροπολογίες του συγητού. Τροπολογία ΦΕΤ 5.019, 5.22, 5.23, 5.24, 25, 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι τροπολογίες αυτές εγκρίνονται. Μετά τροπολογίες FDD που μπορούν να ψηφιστούν μαζί. 56 ο πρόεδρος εφόσον οι τροπολογίες της ΑΦΕΤ ψηφίστηκαν, εγκριθήκαν, αυτές εδώ καταπίπτουν. Και πάμε τώρα σε ξεχωριστές ψηφοφορίες που όμως θα ψηφιστούν τουλάχιστον σε δύο ομάδες Πρώτη ομάδα 8257, 8258, 8259 και 8260. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίστηκαν, εγκρίνονται αυτές τις τροπολογίες. Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, απερίφθησαν. Ζητώ συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Και μετά τροπολογίες ΑΦΕΤ 50-20 και 50-21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται στη γραμμή 200 τροπολογία SER 8210 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται Και τώρα έχουμε τρεις τροπολογίες που θα ψηφιστούν ομαδικά. Η, η BODS 2802 με προφορικές τροπολογίες του εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Άποχες. Οι τροπολογίες αυτές απορρίπτονται. Ερχόμαστε τώρα στο τμήμα 1 δηλαδή προπολογισμό του Κοινοβουλίου πρώτη υποομάδα υπέρ κατά αποχές αυτή η πρώτη υπομάδα εγκρίνεται δεύτερο ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Λοιπόν, οι άλλες τροπολογίες περνάμε αυτές που ψηφίζονται ξεχωριστά. Κύριε Σιγητά, ζητώ συγγνώμη, νομίζω ότι θετήσαμε τα δύο πρώτες ομάδες, δηλαδή κυρώσαμε τις συμβιβασμούς που επετέφθησαν. Μπορούμε να ψηφίσουμε και αυτό εδώ σαν ομάδα ή να τα απορρίψουμε. Η πρότασή σας δεν δημιουργεί καμία αντίρρηση. Συμφωνούμε. Καλώς έχετε τον κατάλογο. Δεν αξίζει το λόγο τώρα να σας το διαβάσω. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ των τροπολογιών που υποτίθεται θα ψηφίζαμε ξεχωριστά. Ευχαριστώ. Ποιοι έχουν αντίρρηση, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τώρα, όσον αφορά τα αποθεματικά, έχουν τρομολογία BOTS 4320 που ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτονται. τελευταίος κατάλογος ψηφοφοριών που είναι οι πληρωμές. Sur les paiements, Έχουμε πρότυπο ομάδα που ψηφίζουμε υπέρ. κατά αποχές αυτή η υποομάδα εγκρίνεται δεύτερη υποομάδα υπέρ κατά άποχες και η δεύτερη υποομάδα εγκρίνεται αυτόνα στις ξεχωριστές ψηφοφορίες πρώτη τροπολογία 7850 υπέρ κατά άποχες απορρίπτωτε, η FTD 7976 υπέρ κατά άποχες απορρίπτωτέ, η FTD 7977 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Βοτς 4110 έχει αποσυρθεί. Τελειώσαμε. Η συνδιαλλαγή ελπίζουμε θα γίνει με την ίδια κατανόηση, διάβια και ειρήνη. Εκεί προσμετρούμε την, ειδική, την ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία των εργασιών μας. Και θα έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε στην ημερήσια διάταξη όσον αφορά τα άλλα θέματα. Πριν από αυτά, ίσως ε, ο εισηγητής θέλει να εκφράσει την ικανοποίησή του. Κύριε Φερναντές, θέλετε να μιλήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η διαδικασία. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους σκιώδης συζητάς, καθώς και τους συντονιστάς των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ βεβαίως τα μέλη της Γραμματείας της ε, Επιτροπής, τους διαφόρους συμβούλους και όλες και όλους τους ε, συμβούλους. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρόεδρε, όλος ιδιαιτέρως. Κατορθώσαμε να συμφιλιώσουμε τις διάφορες ανάγκες, βεβαίως διατηρούμε και την απαραίτητη πειθαρχία. Και χάρη στο συνδυασμό αυτό διαθέτουμε προϋπολογισμό που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Διάφορες προκλήσεις πρόσφατες, όπως για παράδειγμα η κρίση του προσφυγικού που είπαμε εξ αρχής ότι πρόκειται για πολύ σημαντική κρίση και το 1,2 δισεκατομμύρια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει και πόσο επίγουσα είναι η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή, χωρίς βέβαια να λησμονήσουμε και την ανάγκη δημιουργίας απασχολήσεως. Και εκεί η ενίσχυση των διαφόρων προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχολήσεως των νέων και άλλα σχετικά είναι επίσης πολύ σημαντικά. Αναλάβαμε και δεσμεύσεις για προγράμματα που θα υλοποιηθούν μέσα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αυτό που προτείνουμε για τον ορίζοντα 2020 είναι δεσμεύσεις που ήδη είχαν αναλυθεί από πριν και τις οποίες ερχόμεθα τώρα και επιβεβαιώνουμε. Αντιμετωπίζουμε και την κρίση του γάλακτος με έξτρα 500 εκατομμύρια για στήριξη των γαλακτοπαραγωγών Βεβαίω θα πρέπει να δούμε τώρα εάν το Συμβούλιο των Υπουργών όντως θα δώσει συγκεκριμένη μορφή και θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που το ίδιο έχει αναλάβει. Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε την θέση τους. Θα πρέπει να δούμε να υλοποιείται η ελληνική, να γίνεται πραγματικότητα η ελληνική και για το σχέδιο πληρωμών που έχουμε καταστρώσει. Η συνένεση που διαμορφώθηκε εδώ στους κόλπους μας ελπίζω ότι θα βρει ανταπόκριση και στο Συμβούλιο Υπουργών, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δράσει ταχύτατα για να αντιμετωπίσει έκτακτες προκλήσεις. Πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και κάθε ευελιξία που προσφέρει ο προϋπολογισμός μας για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε στις έκτακτες αυτές καταστάσεις. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κονδύλια εκτάκτου χαρακτήρα. Αυτό άλλωστε απαιτούν και οι Ευρωπαίοι πολίτες από εμάς. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πράγματι πρόκειται για εμπνευσμένη ομιλία. Βεβαίως το επόμενο στάδιο θα είναι η συνδιαλλαγή, όπου ελπίζω να δούμε πολλοί αριθμούς τους υπουργούς και να μπορέσει να διεξαχθεί διάλογος ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία των χωρών μελών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους επόμενους μήνες ελπίζω να μπορέσουμε να δούμε και υπουργού εδώ ενώπιόν μας. Πώς θα κάνουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση αν δεν έχουμε άμεση επαφή με τους υπουργού. Βεβαίως έχουμε μέγιστο σεβασμό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως χρειάζεται άμεση επαφή μεταξύ των δύο σκελών της αρχής του προϋπολογισμού, δηλαδή Συμβούλιο Υπουργών και Κοινοβουλίου. Διότι τελείως θα είναι απογοητευτική εξέλιξη. Όταν τα λέμε εδώ μεταξύ μας, ωραία τα πάμε. Ψηφίζουμε και ιδίω δαπάνες εύκολα. Πιο δύσκολα είναι τα πράγματα για τους πόρους. Όταν όμως έρχεται η ώρα της συνδιαλλαγής και ενδεχομένως και του τριμερούς διαλόγου, διότι δεν απέληξε η συνδιαλλαγή μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Θυμούμε και από την πρώτη μου εμπειρία ως Πρόεδρο προέτους η κυρία Γουάρδια Ζαμπάλ είχε υποβάλει τα σχέδιά της με πολύ πειθό αλλά τελικά στην έξοδο δεν μείναν και πολλά πράγματα από αυτά. Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Υπάρχουν στιγμές που προσφέρουν μεγάλη ικανοποίηση, αλλά πρέπει κανείς από αυτές τις στιγμές να λαμβάνει δυνάμεις για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τα δύσκολα που έπονται. Ο κύριος Ντεπρέ, συμφωνώ μαζί σας στην διατύπωση της ελπίδας ότι θα προσέλθουν πολλοί άριθμοι υπουργοί του Συμβουλίου. Δεν θα ήθελα να σας απογοητεύσω, φοβούμαι όμως ότι ίσως οι ελπίδες αυτές να μην πραγματοποιηθούν. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο φίλος μας Χωσέ Φερνάντες για τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού, με βρίσκει σύμφωνο και καλά τα πήγαμε. Ωστόσο έχω μια ανησυχία που θέλω να εκφράσω. Μια ανησυχία για, σχετικά με την Επιτροπή μας. Οι δημοσιονομικές προοπτικές αποτελούν ε, περιοριστικό πλαίσιο και για το Κοινοβούλιο και ειδικότερα για την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εάν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών επιλέγουμε μόνο είτε να αποκαταστήσουμε το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε να κυρώνουμε απλώς τα όσα ζητούν οι άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές δεν θα έχουμε πλέον μεγάλη πολιτική βαρύτητα. Απευθύνω λοιπόν έκθεση στο σύνολο των πολιτικών ομάδων για να προβληματιστούμε σχετικά με τις πολιτικές ευθύνες που επιθυμούμε να λάβουμε στο μέλλον δεν μπορούμε απλώς να είμαστε ένα όργανο που θα κυρώνει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των άλλων αρμοδίων επί της ουσίας κοινοβουλευτικών επιτροπών. Διότι οι αποφάσεις που λάβαμε σήμερα διέπονται νομίζω λίγο πολύ από αυτή τη λογική. Και αυτό με λυπεί βαθέως ο πρόεδρος Αρτουή. Και ως πρόεδρος αλλά και προσωπικά θα σας απαντήσω ότι συμφωνώ με τον Χωσέ Μανουέλ και με τον Ζεράλ Ντεπρέ Νομίζω όμως ότι πάσα Επιτροπή Προϋπολογισμών πρέπει να αποφεύγει και τον εφησυχασμό και μέσα στις πολιτικές ομάδες και στις άλλες επιτροπές και στο Συμβούλιο. Δεν είναι, δεν προσφέρουμε καμιά υπηρεσία στις πολιτικές μας ομάδες αν εφησυχάζουμε. Και θα πρέπει να τη συνοδεύουμε και από την άποψη τη δημοσιονομική. Γιατί είμαστε εκλεγμένοι για να εκπροσωπούμε τους πολίτες. Πώς θα εξηγήσουμε στους πολίτες ότι τα όσα πράττουν εδώ είναι το εφικτό σύμφωνα με τα συμφέροντά τους και ότι σε καμιά περίπτωση δεν επαναπαυόμαστε στα όσα έχουμε επιτύχει ήδη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί δηλαδή η Επιτροπή Προϋπολογισμών να είναι απλώς ο σφραγιδοφύλακας που βάζει τη σφραγίδα και κυρώνει τα όσα έχουν ζητήσει οι άλλοι. Οκ, λοιπόν η συνέχεια θα, τη συνέχεια μόνο θα την παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή. Αν θέλετε να περάσουμε τώρα στο υπαριθμόν 5. Α, με συγχωρείτε, ο κύριο Ρούμπικ του Λαϊκού Κόμματο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω σωστά τοποθετηθήκατε. στον τριμερή διάλογο και στην διαδικασία συνδιαλλαγής θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε ο Υπουργό Οικονομικών τουλάχιστον της χώρας που ασκεί την Προεδρία να είναι παρόν. Να του γράψετε λοιπόν και να του πείτε ότι αναμένουμε να είναι παρόν σε όλες τις διαπραγματεύσεις και να του πούμε ταυτοχρόνως ότι εάν κολλείεται εμείς θα ζητήσουμε αναβολή της ημερομηνία, ημερομηνίας διότι το Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να συζητήσει τα πράγματα αυτά μόνο παρουσία του Προεδρεύοντος. Τότε ας αποφασίσει αυτός εάν θέλει να έρθει ή όχι. Τουλάχιστον με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσουμε την παρουσία του Προεδρεύοντος. Αν δεν έχει χρόνο ο ίδιος, ε, τότε δεν θα έχουμε χρόνο ούτε και εμείς. Νομίζω ότι είναι η μόνη σωστή διαδικασία για να μπορέσουμε να τον φέρουμε στις διαπραγματεύσεις. Με μια παραλλαγή ότι θα πρέπει να προσέξουμε οι διαπραγματεύσεις ή δυνατόν, τη συνδιαλλαγή δηλαδή, να γίνονται εδώ, παροιμήν, στο Κοινοβούλιο. Να κάνει λοιπόν η δική μας διοίκηση όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες και το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να μας υποστηρίξει, ώστε οι διαβουλεύσεις να γίνονται εδώ, σε σωστό πλαίσιο, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως να δείξουμε την απαραίτητη φιλοξενία στο Συμβούλιο Υπουργών. Αν θέλουμε να αποκατασταθεί καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και εφόσον όντως διεξαχθεί η διαβούλευση εδώ, τότε εμείς είμαστε οι κύριοι της διαδικασίας Master of Procedure και μπορούμε να υποδείξουμε και το πού, σε ποια αίθουσα δηλαδή, και το πώς θα γίνει η διαδικασία. Αυτό άλλωστε ενισχύει και τη δική σας θέση ως επικεφαλής του πρωτοκόλου για τη διαδικασία της συνδιαλλαγής. Και έτσι νομίζω θα δείξει το Κοινοβούλιο ότι είμαστε εν τέλει σοβαροί ε, αντισυμβαλόμενοι ή συνομιλητές του Συμβουλίου. Μάλιστα σας ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος. Α, τουί. Κατανοώ απολύτως το έτοιμά σας και το συμμερίζομαι. Από τις 1 Ιουλίου, από τότε που το Λουξεμβούργο ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών, ο Υπουργό Οικονομικών έχει, Λουξεμβούργο Λουξεμβούργου ενώ, έχει φανεί ιδιαίτερα συνεργάσιμος. Διεξήχθη ήδη ένας τριμερής διάλογος όπου συμμετέσχει ο ίδιος τα δε λόγια του ήταν ικανοποιητικά με την έννοια ότι ανέλαβε δεσμεύσεις και ελπίζω πολύ να αποδώσουν καρπούς. Πάντως θα του υπενθυμίσω τις δεσμεύσεις του αυτές. Αν θυμάστε πέρσι είχαμε αποφασίσει να στείλουμε τους συνεργάτες μας, τους βοηθούς μας στην ε, συνδιαλλαγή. μια υπόθεση που δεν πρέπει να λησμονήσουμε υπάρχει και αυτή εάν δηλαδή η εκπροσώπηση του Συμβουλίου Υπουργών είναι σε χαμηλό επίπεδο, υποτιμημένο ας πούμε, τότε και εμείς θα πράξουμε ούτως. Και βεβαίως να μην μου θυμώσουν τώρα οι συνεργάτες μας για αυτό που λέω. Ας δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Γέγκερ για Κάποιος ζητεί το λόγο. Ο κύριο Τάραντ. Πολύ σύντομα. Δεν μπορούμε να στείλουμε τους συνεργάτες μας, διότι δεν αυξήσαμε τους μισθούς τους. Τότε προτιμώ λοιπόν να τηρήσουμε την ε, γαλλική παράδοση της καινής έδρας. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι είναι αφοσιωμένοι στο κοινό συμφέρον οι συνεργάτες μας και ότι κατανοούν ότι περνούμε δύσκολες περιόδους δημοσιονομικά και ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δημόσια οικονομικά της Ευρώπης. Ο Δής επιθυμεί να λάβει το λόγο για τις ψηφοφορίες που έγιναν για τον προϋπολογισμό 2016. Έχουμε άλλους φακέλους που αναμένουν για τις, ε, για την ε, χρήση κονδυλίων του Ταμείου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης. Ιδίω για μια υπόθεση της αυτοκινητοβιομηχανία Opel. Ο κύριο Γκάιερ δεν θέλει να μιλήσει. Έχουμε μια σειρά τροπολογιών. Τροπολογία μόνο 3. Ποιο είναι υπέρ, Μπορούμε να, κάνουμε, να ψηφίσουμε όλες μαζί τις τροπολογίες, λέτε. Υπάρχουν και δύο τροπολογίες της κυρίας Μυριαντά για τις τροπολογίες της Επιτροπής Απασχολήσεως που είναι 7 συνολικά 3 έως 9 όλες μαζί ψήφι υπέρ ευχαριστώ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 2 της κυρίας Μυριάντα, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαρθμονένα, 1, κυρία Μυριάντα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. Επί του συνόλου του κειμένου, ονομαστική ψηφοφορία αυτή τη φορά, Αρχίζει η ψηφοφορία. Κύριε Καμέλα, έχετε προβλήματα. Πέρας της ψηφοφορίας. «23 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, ή μάλλον 7 κατά και 4 αποχές. Πάντοτε για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την Ford Genk, έκθεση Rubik. Έχετε το λόγο κύριε. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησεως να φροντίσει τώρα που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα μεταναστευτικό και προσφυγικό στην Ευρώπη και είναι νέες οι καταστάσεις αυτές, να σκεφτούν, να σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορεί να αναλάβει και νέο καθήκον το Ταμείο προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Βεβαίω για την ψηφοφορία αυτό δεν έχει σχέση που λέω, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε νέε προτάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Ο Πρόεδρο. Η μετανάστευση έχει βέβαια κάποια σχέση με την παγκοσμιοποίηση. Και είναι σημαντικέ οι προκλήσει που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Οι συνθήκε υποδοχή στι διάφορε χώρε, οι μεταβατικέ περίοδοι από τι οποίε και μετά θα μπορούν να εργαστούν ε, τα πρόσωπα αυτά, όλα αυτά πρέπει να αρμονιστούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, πρώτη τροπολογία υπαρθμών τέσσερα Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 5 που καλύπτεται όμως, τότε έρχεται η 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά πολλά μέλη της Επιτροπής δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα χρειαστεί λοιπόν να κάνω επαλήθευση με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 9 λοιπόν αρχίζει υπαριθμόν 9 9 του κ. Αντέλ. Τέλος. Εγκρίνεται 27 υπέρ 4 κατά. Σαφώς όμως δεν ήταν 27 μέλη που σήκωσαν το χέρι πριν. Υπάρχουν 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά μου φαίνεται θα απαγορεύσω τις ταμπλέτες λέει ο πρόεδρος αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά επαλήθευση με ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. 13 υπέρ, 18 κατά και μια αποχή. Υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπαρχουν τρία, Νηριάντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. μόνο ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για το σύνολο του κειμένου ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται με ψήφους 26 υπέρ 6 κατά και μια αποχή. 7, 7, 7 ψήφοι κατά. πάντοτε για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, για την υπόθεση της Αλιτάλια έτοιμα από την Ιταλία, έκθεση της κυρίας Βάνα. Παρατηρήσεις όχι. τροπολογία 3. Περ. Κατά. Ορίστε. C'est bon Traduction Είναι là. Να τα ξαναπώ. Ποιο είναι υπέρ της τροπολογίας 3. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά Να ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εσείς κύριε Καλμελιστή, υπέρ κατά. Άρα 19 ψήφοι υπέρ, 11 κατά, 4 αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία 5. Περνάμε στην 6. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 9 ψήφι πέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 12 ψήφι Μα, να σηκώνετε τα χέρια σας. Παρακαλώ δηλαδή. Ποιοι είναι οι υπέρ της 12. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 26 υπέρ, 6 κατά, μία αποχή. Παρακαλώ. Για το φάκελο. Τουλάχιστον στο δικό μου φάκελο, κύριε Γκρέσλε, δεν έχω τις τροπολογίες. Το κείμενο το έχω, όχι τις τροπολογίες όμως. Ψήφισα δηλαδή τροπολογίες που δεν τις γνώριζα ουσιαστικά καλό θα ήταν να τις είχαμε στο φάκελό μας. Αυτό ήθελα να πω. Πρόεδρος, ξέρετε, από χθε το μεσημέρι δεν κάνουμε κάτι άλλο. Ε, ουσιαστικά ψηφίζουμε τροπολογίες. Ναι, για το φάκελο μιλάει η κυρία Γκρέσλη. Δεν είναι, απαγορεύεται να έχουμε ένα πλήρη φάκελο. Ο πρόεδρος, όλα τα λάβατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λοιπόν, τώρα. Προχωρούμε στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εδώ έχουμε κολλήγες τροπολογίες, ο Σίγητης δεν έχει να προσθέσει τίποτε. Σας τα είπε στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής. Πηγαίνουμε λοιπόν στην παράγραφο 1, τροπολογία 7, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 1α. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές, αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 12, ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 3 τροπολογία 13 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 15 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην παράγραφο 3α νέα τροπολογία 16 ψήφι υπέρ κατά θα ελέγξουμε τροπολογία 16 έρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Κύριε Κόλμελ, είστε υπέρ. Άρα 19 υπέρ, 13 κατά, 2 αποχές. Τροπολογία 17 στην παράγραφο 4, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 στην παράγραφο 4 πάντοτε, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 4α 4α9. Τροπολογία 19 Δύο τμήματα. Ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 5. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται Προπολογία 21 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ονομαστικά λοιπόν ψηφίζουμε. προπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 22 ψήφοι κατά, 11 υπέρ, μία αποχή. Τροπολογία 22 υπέρ. 22 κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 23. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5α νέα. Τροπολογία 25. Ψήφι υπέρ. Τροπολογία 25. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράφος 6. Τροπολογία 27. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε την 27. Ελέγχουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία την τροπολή 27. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17 ήταν οι αντίθετες ψήφοι, 12 υπέρ, 3 αποχές. Τροπολογία 28 ψήφοι υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε και πάλι την τροπολογία 28 αυτή τη φορά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Η τροπολογία αυτή εγκρίνεται 18 ψήφι υπέρ 16 κατά. 28. Πάμε στην 29. Ψήφι υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 29. 18 υπέρ 14 κατά μία αποχή, παράγραφος 6α νέα. Τροπολογία 30. Ψήφι Πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31 στην 6β νέα, παράγραφο ψήφι Πέρ. Κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 22 ψήφοι υπέρ και 11, ε, μάλλον 22 κατά 11 υπέρ. Προπολογία 32 στην παράγραφο 7 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 33 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται να το ελέγξουμε όμως Θα επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, πράγματι, 23 ψήφοι κατά, 24 κατά, 8 υπέρ. Απορρίπτεται λοιπόν τροπολογία 35 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στις ιδεολογικές σκέψεις, το Arta Recitals, τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε παρακαλώ, ονομαστικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Η τροπολογία αυτή απορρίπτεται 19 κατά, 13 υπέρ, 2 αποχές. Τροπολογία 4, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στο σε αλφα νέο τροπολογία 6, ψήφι υπέρ. Κατά, προτιμώ να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 6. Πέρας. Η τροπολογία αυτή εγκρίνεται 21 υπέρ, ψήφι υπέρ, 11 ή 12 με τον κύριο Καλμέλ κατά και τώρα ψηφίζουμε ονομαστικά το σύνολο του κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση 21 ψήφι υπέρ 13 κατά. Περνάμε τώρα στην έκθεση 8α. για το διορθωτικό 6 το 2015 έκθεση την Καρδιά Θάμπαλ. Έχετε παρατηρήσεις πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, δεν έχετε. Νομίζω ότι μπορούμε να... Καλό θα ήταν να ψηφίσουμε ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. 31 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 1 εποχή Εγκρίνεται το κείμενο. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Χολμάιερ. Υπάρχει κάτι άλλο που προηγείται. Α, βέβαια. Οι μεταφορές μεταφορές πιστώσεων λόγω και του τρόπου τον οποίο ψηφίσαμε προηγουμένως. Η κυρία Γκαρδιαθάμπαλ δεν έχει κάποια παρατήρηση για τις ε, μεταφορές πιστώσεων αυτές που απορρέουν από τις ψηφοφορίες όπως ψηφίσαμε δηλαδή την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Ονομαστικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Καλησπέρα στις με 25 ψήφους υπέρ 6 κατά μία αποχή ο διορθωτικός προπολογισμός 6 και τώρα πηγαίνουμε στα λοιπά τμήματα και θα δώσω το λόγο στην κυρία Χολμάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να πω σήμερα. Μία μεταφορά για τον Ευρωπαίο Συνήγορο του Πολίτου. Το αίτημα που μας υποβάλλεται είναι από, τον, τη γραμμή του προϋπολογισμού που προβλέπεται για τις μεταφράσεις να αφαιρεθούν 44.000 και από την γραμμή του προϋπολογισμού για θέματα επικοινωνίας προς τα έξω 31.000, συνολικά 75. Ανταυτού, ο Ευρωπαίος Συνήγορος του Πολίτου επιθυμεί να αναπτυχθούν περαιτέρω ή να μπορούν να αγοραστούν οι υπηρεσίες διαδικτύου. 39.000 και 30.000 για την πρόσληψη προσωπικού. για ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσεως διαδικτύου και γλωσσών. 5.000 ευρώ για δαπάνες ταξιδιών για υποψηφίους που προσέρχονται εδώ για να συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις όταν υπάρχουν και νέες έδρες και θέσεις δηλαδή για το προσωπικό και 1.000 ευρώ για να μπορέσει η συνήγορος του πολίτου να αναπτύξει τις γλωσσικές της δεξιότητες. Δεν μπορεί να πει κανεί όχι σε αυτό, σε αυτή τη μεταφορά. Η συνήγορος του πολίτου είναι ε, θηλυκού γένους η, η κυρία συνήγορος του πολίτου. Για Σας ευχαριστούμε κύριε Χολμάγερ. Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε δηλαδή. Κιόλα. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε την μεσαία διάταξη. Να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας ε, είναι αύριο στις 11 όπου θα έχουμε ακρόαση με την κυρία Γεωργίευα. Προβλεπόταν 7 Οκτωβρίου μια συνεδρίαση, η οποία δεν θα διεξαχθεί, δεν έχει λόγο. Επόμενη συνεδρίαση, Βρυξέλλες, 12 και 13 Οκτωβρίου. Θέλει κανείς το λόγο στα διάφορα Ε, είναι σαφές επίσης ότι δεν έχει συνεδρίες ούτε σήμερα το απόγευμα, ούτε αύριο το πρωί 9 ούτε το απόγευμα, ούτε και την Πέμπτη. Λοιπόν, εδώ κηρύσω τη λήξη της ε, συνεδρίασης. Διακόπτουμε για 10 λεπτά, γιατί έχουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών στις 11. Στις 11. Et ε, voilà.